μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, τους φιλήσατε όλους. Πάμε τώρα. Έχουμε και επεξηγήσεις ψήφου. Mr. Mamikins. Ο κύριος Μαμίκινς. Dear colleagues, dear colleagues, we already... Οι ε, συνάδελφοι, έχουμε περάσει επεξηγήσεις. Παρακαλώ πρέπει να ακούσουμε τους συναδέλφους μας που έχουν επεξηγήσεις ψήφου να κάνουν. Λοιπόν, έχουμε τη σύσταση της κυρίας Καλνιέτε. Συμφωνία πλαίσιο ξενολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Βιετνάμ. Κύριε Μαμίκινς, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Υπήρου μας έδειξε ότι πρέπει να κάνουμε διάφορες αλλαγές σε διάφορες συμφωνίες που έχουμε με άλλες χώρες για να καλύψουμε τη διεύρυνση. Ε, εν αυτό αφορά την... Σε ό,τι αφορά τώρα τις σχέσεις Κροατίας-Βιετνάμ υπάρχουν σε επίσημο επίπεδο εδώ και μία εικοσαετία αλλά δεν έχει καμία από τις δύο χώρες μόνιμη και διαρκή ε, εκπροσώπηση πρεσβεία στην άλλη χώρα. Ωστόσο, σχέσεις έχουν επί μία εικοσαετία και πλέον. Συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, κατάργηση ε, θεωρήσεων για διπλωματικά διαβατήρια κτλ. Από τότε που μπήκε η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμφωνία αυτή πλαίσιο θα δώσει αρκετή ευημερία Ευχαριστώ πολύ και προχωρούμε στη ε, επόμενη έκθεση Μπίλερ πάλι, κύριος Μαμίκινς, πάλι για το Βιετνάμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η Συμφωνία Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ έχει ως βασικό στόχο την προώθηση περαιτέρω εξελίξεων και τη δυναμική στι αμοιβέ μας σχέσεις σε διάφορου τομεί Θα προωθηθούν οι οικονομικές συνεργασίες, ο τουρισμός, οι επενδύσεις με αμοιβαίο σεβασμό των παραδόσεων και των ηθών και των εθήμων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Όλα αυτά συνιστούν τα θεμέλια των σχέσεων μας με το Βιετνάμ. Ε, είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες, αναδυόμενες οικονομίες στην νοτιοανατολική Αφρική, το Βιετνάμ και στον ειρηνικό γενικότερα. Ε, η προώθηση της συνεργασίας είναι εκ των όνου κάνευ και είναι λογικό βήμα πρόοδου. Άλλωστε, σας ευχαριστώ. Yes, it works. Πρέπει να σταματήσουμε εδώ να βγάζουμε λόγους κατά των τρίτων χωρών και να τους λέμε τι να κάνουν και πώς συμπεριφέρονται. Αναφέρομαι όλος ιδιαιτέρως στο κείμενο της παραγράφου 33 της εκθέσεως. Μιλάμε στο Βιετνάμ. Του λέμε τις για τις θεωρήσεις και πού πρέπει να έχει επιγραφές η πρεσβεία. Αυτά είναι ανοησίες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι τρίτες χώρες έχουν δική τους δημοκρατική ζωή, έχουν κυριαρχία. Και το λέω γενικά, σαν θέμα αρχής. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά εδώ πέρα. Υπερβολικά συχνά. Και πρέπει να σταματήσουμε να επιβάλλουμε τη δική μα νοοτροπία σε άλλους λαού του κόσμου. Ευχαριστώ, Πολτσάκ. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Πόλτσακ, που μου δίνετε το λόγο. Συμμετείχα στη συζήτηση για το Βιετνάμ και δεν γνώριζα τα άρθρα 33 μέχρι 35 λεπτόμερος. Τα διάβασα τώρα και δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην ε, στηρίξω τη συμφωνία. Οι απαιτήσει ε, που ε, έχουμε επιβάλει ήταν λογικές άρθρα 34 μέχρι 35 στη Συμφωνία Πλαίσιο. Τίποτα το εξαιρετικό και το έκτακτο και το ασύνηθες. Υπερψήφισα και πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθεί στατηγικέ σχέσεις με την Νοτιοτελική Ασία. Είναι σημαντικό αυτό για περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων και ευχαριστώ. Ε, Προχωράμε λοιπόν. Και πάμε στην πρόταση ψηφίσματος για την Νομισματική Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την ε, ενοποίηση την κοινό νόμισμα στην Ευρώπη. Οδήγησε σε μεγάλη κρίση και οδήγησε σε πολιτική αποσυναρμολόγηση της συνεργασίας μας. Θα θέλαμε λοιπόν να αποσυρθούμε από την πολιτική, γιατί θα έπρεπε να είμαστε λογικοί, αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την κρίση αυτή και να μην τη χρησιμοποιήσουμε ως πρόσχημα για να στερήσουμε από τα κράτη-μέλη τμήματα της εθνικής τους κυριαρχίας. Ε, θα πρέπει ε, να ε, λάβουμε υπόψη τη Βρετανική θέση. Ε, Δυστυχώ είναι απόδειξη σημαντική πολιτική ανευθυνότητα, ε, προσπαθώντα υποτίθεται ε, να εξυπηρετήσει του λαού. Αλλά είναι θέμα επιλογή και εμεί επιλέγουμε την εθνική μα κοινωνία. Σα ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το σύστημα του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου ε, ίσχυε πλέον πέντε χρόνια και επηρεάζει την άσκηση τη πολιτική, στον οικονομικό τομέα σε ό,τι αφορά και το θέμα τα συντονισμού ε, στα τα κράτη-μέλη. Τα εθνικά συστήματα και τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, περιλαμβάνει ελέγχους σε επίπεδο εφαρμογής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί τέτοιου ε, ελέγχου στα εθνικά συστήματα. Πιστεύουμε όμω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει σε μεγαλύτερο βαθμό, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, να υπάρχει μεγαλύτερο έλεγχο τη ε, διαχείρισης. Και αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με το Κοινοβούλιο όταν προετοιμάζει τη Λευκή Βίβλο για την Ένωση Εποπτείας και σε ό,τι αφορά το πρώτο και το δεύτερο αυτό έτος. Ε, επικεντρωνόμαστε πιο πολύ σε τρίτο και τέταρτο κομμάτι και αυτό το υποστηρίζω. Let me take you back to Άρνοντ, θα ήθελα να σας ε, θυμίσω ότι η δεκαετία του 90, όταν ε, ο Βρετανός Τζον Μέιτζορ πρότεινε ένα ευρωπαϊκό κοινωνόμισμα, αυτό τότε ήταν μια καινούργια ιδέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά ε, μπήκαμε στο μηχανισμό συναλλαγματικής ισοτιμίας σε ό,τι αφορά το συντονισμό της νομισματικής πολιτικής και της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι ε, επλήχθησαν πιο πολύ από ποτέ οι βρετανικές ε, επιχειρήσεις και μας πήρε πάρα πολλά χρόνια να ανακάμψουμε. Ευτυχώς που δεν μπήκαμε στο ευρώ. Το ίδιο μπορεί να είχαμε λουστεί. Όπως ε, πολλές χώρες που μπήκαν σε αυτή την νομισματική ένωση. Ο κύριος Μέιτζορ σύστησε λοιπόν τότε Ευρωπαϊκή, το Ηνωμένο Βασίλειο να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω ότι έκανε και πάλι λάθος. Περνάμε τώρα στην ε, έκθεση του κυρίου Πρέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ετήσια έκθεση του 2014. κυρία Ζάμπορσκα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πρόεδρο, φέρει μια μεγάλη ευθύνη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ε, ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, σε ό,τι αφορά το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και θα πρέπει επίσης ε, να βρήκε τρόπους αποτροπής των μεταναστευτικών ροών από χώρες όπου όμως δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ισορροπημένο το κείμενο και σε ό,τι αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής. Ε, είναι σωστά τα όσα επισημαίνονται. Εκ παράλληλη, το κείμενο περιλαμβάνει τροπολογίες που ξεπερνούν τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία τα ανθρώπινα δικαιώματα για να προβληθούν επιχειρήματα υπέρ των αγλώσεων και των γάμων ομοφυλόφιλων. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάστηκα να καταψηφίσω την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ μερικές χώρες αναπτύσσουν ε, τις επαφές τους, άλλες ε, εγκλωβίζονται σε στενά συμφέροντα. Νομίζω ότι είναι χρέος και καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να υπερασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να ξεχνάμε και την ιδιαίτερη πορεία που ακολουθεί κάθε χώρα. Και αν μιλούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως οικουμενικό αγαθό, δεν θα πρέπει παρόλα αυτά να ξεχνούμε ότι ο, ίσως ο καθένας τα αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο. Ο καθένας θα πρέπει με το δικό του τρόπο να προωθεί τα δικαιώματα και τις αξίες, τηρώντας βέβαια και σεβόμενος και τα δικαιώματα και τις αξίες των άλλων. Γενικώ ε, υπερψήφισε την έκθεση πάντω. Üdvözlöm, hogy a jelentés az unió belső és külső ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην έκθεση λοιπόν αυτή το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να δείξουμε μία συνέπεια μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστούμε λοιπόν την προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής. Η εξωτερική πολιτική σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, αποτελεσματική. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να μιλήσω για τις αυτόχθονε μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συχνά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί κριτική κατά τρίτων χωρών για παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αλλά οι μειονότητες ε, στην, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 10% του πληθυσμού και δεν ε, τις προσέχουμε όσο θα έπρεπε. Όλοι υποστηρίζουμε λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αυτή η έκθεση δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα μιλούν με μία και μόνη φωνή για τέτοια θέματα. Μία μόνη φωνή. Αυτό πώς συνάδει με τα κυριαρχά δικαιώματα των κρατών για εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα αναφέρομαι στις τροπολογίες που εγκρίθηκαν σήμερα σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή, σε ό,τι αφορά τον ορισμό ενός νέου είδους ε, πρόσφυγα, του πρόσφυγα λόγω κλιματικών ε, ε, συνθήκων. Κατά δεύτερον, τα συστήματα ποσοστώσεων. Αυτά είναι για τις γυναίκες, για την δημοκρατία, στην, στις επιχειρήσεις. Πώς Α, πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτές οι τροπιαστικές ποσοστώσεις είναι καλές και πώς μπορούμε, θεωρούμε να τα επιβάλλουμε εκτός της Ευρώπης. Είναι πραγματικά παράλογο. Και τρίτον, είμαι προσωπικά κατά κατά της θανατικής ποινή, αλλά δεν είναι στο χέρι μας και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να κάνουμε μάθημα στους άλλους ότι δεν τι θα πρέπει να κάνουν. Είναι θέμα των κυριάρχων κρατών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, την 20η επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Dayton, ο κύριος Μάε Μίκινς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Dayton, κάτι που έφερε στα Βαλκάνια την πολυπόθητη ειρήνη και έθεσε τις βάσεις, ε, υποτίθεται, για μια δημοκρατική κοινωνία και δημοκρατία στη Βοσνία και Ζεγοβίνη. Δυστυχώς όμως η αρχή της συνένεσης που χρησιμοποιήθηκε στη Συμφωνία του Ντέιτο δεν έλυσε τα προβλήματα των εθνοτικών διαφορών. Η Βοσνία και Ζεγοβίνη εξακολουθεί να είναι μια διχασμένη χώρα και συνεχίζουν οι διαφορές μεταξύ των κοινοτήτων, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην κυβέρνηση. Μάλιστα η Ρεπούμπλικα Σέρψκα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του διαχωρισμού που υπάρχει μεταξύ των κοινοτήτων. Δεν είναι δυστυχώς ακόμη αρκετά καλές σχέσεις ε, μεταξύ τους. Πάντως θα πρέπει να στηρίζουμε συνεχώς την ειρηνευτική διαδικασία. Ευχαριστώ. Έκθεση Βαλέρο, κύριε Μάμικινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα νομικά δεσμευτικό σύστημα στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούμε εμπόριο συμβατικών όπλων με τους διάφορους παγκόσμιους εταίρους μας. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι ευρωπαϊκές χώρες είναι στις πρώτες θέσεις σε αυτό το τομέα. Εξάγουμε όπλα σε πολύ μεγάλους αριθμούς ε, για εκατομμύρια ευρώ. Αλλά χρειάζεται ομοιόμορφη νομοθεσία για το εμπόριο αυτό. Βέβαια, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αναπτύξει την πολιτική της, η οποία όμως θα πρέπει να είναι σύμμορφη με τα, η οποία μάλλον είναι σύμμορφη με τα συμφέροντά της, όμως το εμπόριο αυτό θα πρέπει να γίνεται με διαφανή τρόπο και οποιαδήποτε παράβαση αυτών των νομοθεσιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα. Ο κύριος Σόγκορ. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν τα θέματα σε ό,τι αφορά την κυριαρχία των, Ευρωπα... Ε, κρατών μελών. Η έκθεση λοιπόν κατηγορεί τα κρατημέλη και ασκεί κριτική κατά των κρατών μελών γιατί δεν τηρούν αυτές τις κοινέ τοποθετήσεις και ε, εφαρμόζουν πολλές κυρώσεις. Αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο τομέα όπου τα κράτη-μέλη ποτέ δεν θα παραδώσουν, θα εκχωρήσουν τις αρμοδιότητές τους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις εξαγωγές των όπουλων των κρατών μελών θα πρέπει να δούμε κατά πόσον συνάδουν αυτοί, αυτές οι πολιτικές με τους ε, ε, στόχους της εξωτερικής πολιτικής. Και εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση. Οι εξαγωγές όπλων των κρατών μελών υπονομεύουν τις κοινέ μας αρχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα επιθετικής ποικιλία. Ο κύριος Μαμίκινς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για 17 ολόκληρα χρόνια ισχύει η σχετική οδηγία που προβλέπει εξαίρεση από την κατοχήρωση με διπλώματα ευρυστεχνίας ε, των φυτικών γνωρισμάτων και των ε, ε, βελτιώσεων φυτών που είναι συνέπεια μιας ουσιαδός βιολογικής διεργασίας. Δυστυχώς, το Μάρτιο του 2015 το διευρυμένο γραφείο προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία ε, περιφρόνησε αυτή την οδηγία και κατέληξε στην απόφαση ότι οι ντομάτες και τα μπρόκολα μπορούν να κατοχυρωθούν με διπλώματα ευρεσιτεχνία, συγκεκριμένε φυτικέ ποικιλίε. Δημιουργεί έτσι ένα πολύ αρνητικό δεδικασμένο και προηγούμενο για δυνατότητα κατοχύρωση με διπλώματα ευρεσιτεχνίας κάποιων φυτικών ε, ποικιλιών ε, φρούτων και λαχανικών θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να επανέλθει στο σωστό δρόμο το Γραφείο Ευρεσιτεχνία. Η κυρία Χάρκιν, εγώ με ιδιαίτερη χαρά υπερψήφισα το ψήφισμα γιατί είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε την εξαίρεση για τους βελτιωτές. Δηλαδή να έχουν πρόσβαση οι καλλιεργητές σε όλο το βελτιωτικό υλικό. Όλοι μάλιστα οι βελτιωτές. Και αυτό ισχύει για τις φυτικές ποικιλίε αλλά και για τις ε, φυλές των ζώων θα πρέπει οι ποικιλίε αυτές να είναι ε, προσιτές σε όλους όσους θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν για βελτίωση και να μην κατοχυρώνονται από δίπλωμα επιστεχνίας. Αυτό ισχύει για τους καλλιεργητές, για τους κυπουρούς, για τους γεωργούς, για όλους τους ενδιαφερόμενους. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογή και την ε, ερμηνεία της οδηγίας 44 ε, του 98 γιατί είναι απαράδεκτο προϊόντα που αποτελούν συνέπεια ουσιοδός βιολογικών διεργασιών να κατοχυρώνονται από δίπλωμα ευρυστεχνίας. Θα πρέπει να εμείνουμε στην εξαίρεση των βελτιωτών, δηλαδή να επιτρέπεται η ελεύθερη συναλλογή τέτοιου γενετικού υλικού. Και λυπούμε για μία παράγραφο που τελευταία στιγμή προσθέθηκε στο ψήφισμα που κατά τελειπού είναι πολύ σωστό. Επόμενο θέμα, η κατάσταση στο Μπουρούντι. Ο κύριος Μαμίκινς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για πολλούς και διάφορους λόγους, οι αφρικανικές χώρες είναι αυτές οι οποίες, αν και έχουν ανακτήσει την ανεξαρτησία τους, εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες λόγω ε, φτώχεια, σε παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. λοιπά και και λόγω σαθρών δομών. Ορισμένε χώρε τα καταφέρνουν καλύτερα. Ε, όμως το Μπουρούντι είναι μια από τι πιο προβληματικέ χώρε, παρότι έχει κερδίσει την εξαρτησία του εδώ και αρκετά χρόνια. Η εθνική κάθαρση, το γενοκτονία, οι εμφύλοι πόλεμοι, πολύ μεγάλη φτώχεια και πολύ αδύναμη κατάσταση όσον αφορά την παιδεία και την υγεία. Πράγματα τα οποία οδήγησαν σε βάθηση της κρίσης. Προστασία του Εθνικού Πάρκου Βερούγκα στην Δημοκρατία του Κονγκό. Ο κύριος Μαμίκινς. Το εθνικό, ο Εθνικός Δρυμός Βιρούγκα είναι ένα από τους παλαιότερους στην Αφρικανική Ήπειρο και είναι εξαιρετικά πλούσιο σε βιοπικιλότητα και σε διάφορα ζωικά είδη. Δυστυχώς από τότε που μπήκε στον κατάλογο της ε, παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO απειλείται διαρκώς. Η τοπική κυβέρνηση έχει ε, ε, δώσει ε, δικαιώματα εξόρυξης πετρελαίου σε διάφορες εταιρείες και στην Κεντρική Αφρική υπάρχουν διάφορες ε, ματηρές σειράξεις. Ε, επίσης γίνεται παράνομη λαθρο, λαθροθυρία ζώων, αγρίων ζώων. 140 φύλακες του Δρυμού έχουν χάσει τη ζωή τους τα περασμένα χρόνια και εγώ είμαι πολύ περήφανος που ως Κοινοβούλιο προσπαθούμε να στηρίξουμε τη διατήρηση αυτού του Δρυμού και γι' αυτό υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης ε, θα σας ταλούν προς έγκριση στην αρχή της επόμενης συνόδου. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις... Ε, τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν σήμερα θα διαβιβαστούν